έληξε η περίοδο συνόδου αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσοι δεν έρθετε στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, καλές διακοπές. Έληξε συνεδρίαση.